Φίλε, ναι, δεν νομίζω ότι θα προσθέσουν πολλά μέλη στη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Απασχόλησης, γιατί ε, πολλοί συνάδελφοι ε, έχουν πάρα πολλά να κάνουν στο τέλος της ολοκλήρωσης, δηλαδή της βουλευτικής τους ε, θητείας και της προετοιμασίας των εκλογών. το καθεστώς διαρμηνίας για τη σημερινή συνεδρίαση είναι ότι εκτός από τα μαλτέζικα και τα κροατικά έχουμε πλήρες καθεστώς διερμηνία σε όλες τις γλώσσες. Περνάμε στο σημείο 3 της ημερήσιας διάταξης, έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων συγκεκριμένα της 26 Φεβρουαρίου του 2019. Μπορούμε να εγκρίνουμε λοιπόν αυτά τα πρακτικά. Θεωρούνται ως εγκεκριμένα. Περνάμε στο σημείο 4 της ημερήσιας διάταξης και αυτό είναι η ενημέρωση σχετικά με τις τρέχουσες διοργανικές διαπραγματεύσεις και καθώς ο κύριος ε, ε, Μπάλα σε βιάζεται και θα πρέπει να αποχωρήσει, χαίρομαι που είναι στην ώρα του εδώ έτσι ώστε να μας ενημερώσει σύντομα. Και αύριο όταν θα κάνουμε την ε, πέμπτη, τον πέμπτη τρίμερη διάλογο για αυτό το ζήτημα, να ξέρουμε τι ακριβώ θα συζητηθεί. Κύριε Μπάλα, λοιπόν, έχετε το λόγο για να μα εξηγήσετε τι ακριβώ συμβαίνει εκεί. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε θα συνημερώσω για αυτό το τριμερή διάλογο. Ένα τρίλογο λοιπόν, ο οποίος ίσως θα είναι ο τελευταίος. Οπωσδήποτε θα είναι ο τελευταίος. Και δεν έχουμε επιτύχει συμφωνία ακόμα, ε, ελπιστούμε ότι θα έχουμε. Αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Θα τα πω πολύ γρήγορα. Το Κοινοβούλιο έκανε πολλές ε, παραχωρήσεις η διαπραγματευτική ομάδα πραγματικά θεώρησε ότι έπρεπε να το κάνει για να προχωρήσουμε. Το Συμβούλιο όμως δεν μετακινήθηκε πολύ από τη θέση του. Ούτε μία φορά δεν έκανε κάποια κίνηση. Απλώς ε, έκανε κάποιες προσπάθειες σε ορισμένα θέματα. Τρία ζητήματα όμως πρέπει να επιβεβαιωθούν σήμερα. Πρώτον, η ικανότητα των κρατών μελών να κρίνουν εάν δεν υπάρχουν απαντήσεις ή ανεπαρκείς στις ερωτήσεις όσον αφορά την εφαρμοστέα ε, νομοθεσία. Υπάρχει επίσης το θέμα των διασυνοριακών εργαζομένων. Τώρα η Κομισιόν κυρίως αρχίζει να κάνει κάποιες προτάσεις οι οποίες φαίνονται αρκετά ενδιαφέρουσες αλλά δεν έχουν ακόμα συζητηθεί στην τελική τους μορφή με το Συμβούλιο. Ε, επίσης, πολυδραστηριότητα. Ε, που εργαζόμενοι σε πολλούς ε, κλάδους ή σε πολλές χώρες, ποια είναι τα κριτήρια ε, βάσει των οποίων θα κριθεί που θα ανήκουν όσον αφορά την κοινωνική ασφάλιση. Προς ώρα το Συμβούλιο, όπως και η Επιτροπή άλλωστε, δεν δέχεται κανένα κριτήριο το οποίο θα συνδέεται με την κατάσταση του εργαζομένου, δηλαδή που εργάζεται πραγματικά. Εμείς πιστεύουμε ότι θα υπάρξει, πρέπει να υπάρχει το, το κριτήριο αυτό, όπως άλλωστε θα πρέπει να υπάρχει και το κριτήριο της επιχείρησης. Δεν έχουμε προχωρήσει λοιπόν. Όσον αφορά τα υπόλοιπα, που είναι πολλοί τομεί, έχουμε προχωρήσει πολύ και θα ήταν πραγματικά κρίμα, ειλικρινά το λέω, θα ήταν κρίμα εάν ε, σε αυτό το σημείο και παρά τις πρόοδους που έχουμε ήδη κάνει αλλού ε, τελικά να αποτύχουμε και να μην έχουμε συμφωνία. Ευελπιστούμε ότι αύριο θα τα καταφέρουμε. Thank you, Mr. Ballas. Perhaps have... Ευχαριστούμε. Ε, κύριε Μπάλας, έχουμε ένα-δυο λεπτά ακόμα στη διάθεσή μας αν υπάρχει κάποιο ερώτημα από κάποιο συνάδελφο. Δεν βλέπω να ζητάει όμως κανείς το λόγο, οπότε είμαστε ικανοποιημένοι από αυτή την ενημέρωση από την πλευρά του κυρίου Μπάλλα. Και ε, ο επόμενο λοιπόν τριμερή διάλογο θα λάβει χώρα αύριο. Οπότε φαντάζομαι, κύριε Μπάλλα, και η αντιπροσωπεία μας θα μπορεί να μας πει κατά πόσο είναι πράγματι δυνατό να συνεχιστούν και άλλες συναντήσεις, να συνεχίσουμε δηλαδή και με άλλους τριμερείς διαλόγους ή οτιδήποτε άλλο, προκειμένου να ε, προσπαθήσουμε να φτάσουμε σε μια λύση ή να μας πει αντιθέτως εάν θεωρείται ότι πλέον δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί περαιτέρω πρόοδος. Δεν ξέρω τι νομίζετε ότι θα συμβεί κύριε Μπαρασάβε. Ναι, νομίζω ότι μπορούμε ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε. Αύριο είμαι σίγουρη ότι θα υπάρξει συμφωνία. Στην τελευταία τριμερή διάλογο ήμουνα σίγουρη ότι όλα είχαν σταματήσει και δεν θα υπήρχε συμφωνία. Αλλά εξελίχθηκαν τα πράγματα. Θα δούμε αύριο. Συνεχίζεται η ιστορία αυτή. Και εγώ την ίδια εκτίμηση είχα ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. τις δύο προηγούμενες συναντήσεις, αλλά θα δούμε πραγματικά και από την άλλη πλευρά και από την να καταλήξουμε σε μια κάποια συμφωνία. Σας ευχαριστώ για την παρουσίαση αυτής της έκθεσης και σας ευχαριστώ που παθήσατε μαζί στις δώσετε προφορίες πριν αρχίσει η σημερινή συνεδρίαση. Τώρα, η αυριανή συνεδρίαση, συγγνώμη. Τώρα. το σημείο 5 της ημερήσιας διάταξης που αφορά τη συμφωνίες συμφωνίας στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου και, και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει αναβληθεί για αργότερα το θέμα αυτό. Δεν σας προκαλεί καμία κατάπληξη φαντάζομαι. Πρόκειται για μια πάρα πολύ κρίσιμη στιγμή το θέμα αυτό και θα επανέλθουμε βεβαίως. Περνάμε στο σημείο 6 τώρα. Κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Μητροφάνο, ο οποίος είναι ο εισηγητής υπεύθυνος για την έκθεση αυτή. Κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ε, σκιώδεις εισηγητές για την πολύ παραγωγική θετική εργασία που κάναμε για το θέμα αυτών των κατερνίων γραμμών. Ενέκρινε την πρόταση σε απόφαση του Συμβουλίου η Επιτροπή για την πολιτική απασχόληση των κρατών μελών και διευθυντηρίες γραμμές οι οποίες ισχύουν όπως ξέρουμε, καταρχάς το 2011. Όπως σας είπα και προηγουμένως, σας είπα ποια ήταν ε, η πορεία των διαπραγματεύσεων ε, με το Συμβούλιο και ήταν πολύ δυναμική προορατική η Βουλγαρική Προεδρία, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω για την στενότερη συνεργασία μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου για την προετοιμασία του τελικού κειμένου. Θα πρέπει όμως να αποδεχθούμε το ότι Υπήρχαν κάποια θέματα που πρόκειψαν κάτι τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και μπλοκαρίστηκαν κάποια σημεία εκ μέρους του Συμβουλίου και εξαφανίστηκαν. Κατά τη διάρκεια της ε, διαδικασίας διαπραγμάτευσης και της ομάδας εργασίας για τη διάρκεια της και πρέπει να πω ότι περασπίστηκαν τι θέσει μα ώστε να ληφθούν υπόψη οι θέσει μας για τη διάρκεια τη τελική απόφαση του Συμβουλίου. Το Συμβούλιο τελικά το μόνο που κάνει είναι να, πρέπει να κάνει είναι να ζητήσει την γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Υπάρχουν κάποια προβλήματα όσον αφορά το τεχνικό κείμενο. Αυτές οι διαπραγματεύσεις θεωρώ ότι όμως δημιούργησαν προηγούμενο και ευτυχώς είναι καλό παράδειγμα της πρακτικής για το μέλλον. Όχι μόνο οι τροπολογίες μας πέρασαν, αλλά κάποιες άλλες δεν πέρασαν και υπάρχει και το θετικό, υπάρχει και το αρνητικό. Σε κάποια σημεία δεν υπάρχει καθόλου πρόεδρο. Λαμβάνοντα υπόψη λοιπόν αυτά που ελέγχθηκαν, σύμφωνα με την απλοποιημένη δικτύα, σύμφωνα με τον ε, ε άρθρο 51, ακολουθούμε την πρόταση την οποία έχει υποβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα δώσω τώρα το λόγο στους κύριους συζητητές. Καταρχήν τον κύριο Μπέγκα εκ μέρους του ΕΛΚ. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Έτσι όπως αντιλαμβανόμαστε εμείς τα πράγματα, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής χαίρει επίσης μιας ε, θετική ε, στάση από το Συμβούλιο και γνωρίζοντα από ε, τα βασικά στοιχεία του κοινωνικού πυλώνα είχαν ήδη εφαρμοστεί σε ικανοποιητικό βαθμό μέσα σε αυτή την πρόταση, θεωρούμε πως αποτελεί τώρα λογική συνέπεια του να ακολουθήσουμε αυτή την προτινόμενη άγουσα με την ε, ταχεία διαδικασία, το fast track procedure, έτσι ώστε τελικά να οδηγηθούμε ε, σε, εκείνο, σε όλα όσα εκείνα ε, θεωρούσαμε εμεί σημαντικά ω Επιτροπή Απασχόληση, δηλαδή μεταρρύθμιση των αγορών εργασία, δημιουργία των θέσεων εργασία, διαβίου μάθηση, ε, επαγγελματικά προσόντα και ούτω καθεξής. Θεω, μπορώ λοιπόν να πω ε, εκ μέρου του ΕΛΚ ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε με αυτή τη διαδικασία και θα την υπερψηφίσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Μπέκερ. Και ε, τώρα ο κύριο Ντέτσνερ ως σκιώδη ηγητή από την πλευρά των σοσιαλιστών. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε είναι μια καλή ευκαιρία να συζητήσουμε αυτή την πρόταση της Ρουμανικής Προεδρίας του Ιουνίου του 2018. Ε, ε, ως θετικό στοιχείο θεωρώ ε, πως το ε, Συμβούλιο τώρα από αποφάσισε να λάβει υπόψη και να επαγχωρήσει έναντι ε, της ε, άποψης ή της γνώμης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την οποία έχει υποστηρίξει εδώ ε, και πολύ καιρό. Δηλαδή μέσα στην νέα πρόταση υπάρχουν σημαντικά στοιχεία αυτής της θέσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και υπάρχουν και συγκεκριμένες κατευθυντήρες γραμμές σε ό,τι αφορά τις συστάσεις αναχώρα που αποτελούσαν και, το, και τμήμα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Ο στόχος είναι να έχουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο συντονισμό των σχετικών δημοσιονομικών εργασιακών ε, και άλλων πολιτικών που σχετίζονται με την απασχόληση και νομίζω πως θα πρέπει να αποτελέσει κάτι που ενδιαφέρει τους πάντες να αποτελέσουμε δηλαδή σημαντικό παράγοντα σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση των περαιτέρω κατευθυντηρίων ε, γραμμών σε αυτό το τομέα. Ε, από την πλευρά δηλαδή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τώρα, πέραν των ε, ζητημάτων επί τη διαδικασία, θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα-δύο σημεία επί του περιεχομένου του ίδιου του κειμένου. Καταρχήν, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε ταχθεί υπέρ τη ε, Περισσότερη ευθυγράμμισης, ε, ε, πιο αυξημένη αν θέλετε ευθυγράμμιση αυτών των κατευθυντήριων γραμμών με τα όσα είχα αποκύψει από το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Η στάση όμως αυτή του Κοινοβουλίου είχε αγνοηθεί από το Συμβούλιο, ωστόσο αποφασίστηκε πως την περίοδο 2020 2021 αυτό θα γίνει. Και το δεύτερο στοιχείο που θα ήθελα να αναφέρω είναι ότι δεν μπορούμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση με τη δική μας ευημερία να επιτρέπουμε την ένδια από την οποία αποφέρουν τα παιδιά. Δηλαδή η παιδική φτώχεια δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί όπω άλλα ε, φτώχεια. Και γι' αυτό εμεί ε, συζητήσαμε να υπάρξουν συγκεκριμένα στοιχεία εδώ που θίγουν την ένδια των ε, παιδιών, αλλά το Συμβούλιο και πάλι δεν είχε συμφωνήσει. Τα παιδιά δηλαδή που διαβιούν σε συνθήκε φτώχεια θα πρέπει να έχουν πρόσβαση χωρί χρέωση ε, υποδομές ε, και υπηρεσίας ε, φροντίδας, κατοικίας, φροντίδα παιδιών, εκπαίδευση και ούτω καθεξής. Η δική μα πρόταση είναι λοιπόν στο μέλλον τουλάχιστον το Συμβουλίο να συμπεριλάβει και αυτό το στοιχείο τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μέσα στο κείμενο. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρο. Υπάρχει κάποιο εδώ που μπορεί να εκπροσωπήσει το ECR. Εάν όχι, να ρωτήσω αν υπάρχει κάποιο εκ μέρου των φιλελευθέρων τη Άλντε. Και πάλι δεν υπάρχει κανείς. Υπάρχει κανείς ε, τώρα από την πλευρά της NGL, Όχι και πάλι. Υπάρχει κανείς από την πλευρά του FDD. Όχι και πάλι. Και υπάρχει κανείς που εκπροσωπεί το ENF. Όχι. Τότε θα δώσω και πάλι το λόγο στον κύριο Μητροφάνοφ, τον εισηγητή δηλαδή. Ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι για τις παρατηρήσεις σας και για την υποστήριξή σας. Νομίζω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να πούμε στους ψηφοφόρους μας ότι κάναμε ένα μεγάλο βήμα προς την κατεύθυνση της κοινωνικής Ευρώπης με την έγκριση αυτής της έκθεσης. Γι' αυτό σας ευχαριστώ πολύ. Θέλω να επαναλάβω απλώς ότι συμφωνώ ε, να προχωρήσουμε, δηλαδή με την πρόταση να προχωρήσουμε με απλουστευμένη διαδικασία και χωρίς τροπολογίες. Λοιπόν, ε, βλέπω ότι υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι. Ε, επομένως, όποιος θέλει μπορεί να ζητήσει το λόγο, Κύριο κύριος Μάνα. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Θεωρώ θετικό το γεγονός ότι βλέπουμε να υπάρχει συνένεση μεταξύ των παριστάμενων ευρωβουλευτών αυτό νομίζω πως καταδεικνύει την ανάγκη του, α, της ύπαρξης κάποιων κατευθυντήριων γραμμών οι οποίες ε, θα γίνουν δεκτούς, ε, ε, αποδεκτές από όλους. Ε, βέβαια είναι σημαντικό πράγματι, όπως το ανέφερε και η Πρόεδρος, ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο ε, προεκλογική, αλλά παρόλα αυτά βλέπουμε για πρώτη φορά το Συμβούλιο να έχει αντιληφθεί ότι είναι σοβαρό το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, μέσα σε αυτό. Δηλαδή, αναφέρεται εκεί σε αριστερέ γραμμέ το τι δεν έχουν κάνει τα κράτη-μέλη ακόμα και τι θα πρέπει να κάνουν από εδώ και στο εξή. Άρα λοιπόν αυτό ακριβώ καταδεικνύει ότι λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη μα το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και ότι οι σχετικέ κατευθυντήριε γραμμέ έχουν να παίξουν σοβαρό ρόλο στο πλαίσιο αυτού του Ευρωπαϊκού Εξαμεινού. Και ένα ακόμα που θα ήθελα να πω είναι ότι ε, ο, ο πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων ήταν κάτι που είχε, ε, ε, στο οποίο είχε ασκηθεί ιδιαίτερη κριτική. Πολλοί είχαν πει δηλαδή ότι αρχίσουμε να παρεμβαίνουμε στον, ε, στον τομέα τη αρμοδιότητα των κρατών μενών, ενώ άλλοι έλεγαν ότι δεν πάμε αρκετά μακριά με αυτόν τον πυλώνα. Βλέπουμε τώρα να υπάρχει ένα κάποιο συμβιβασμό και θα πρέπει να διασφαλίσουμε ε, την εφαρμογή στην πράξη αυτών των δικαιωμάτων που αναφέραμε σας στον πυλώνα με πολύ συγκεκριμένα μέτρα. Αλλά στο πλαίσιο αυτή τη διαδικασία θα πρέπει να εμπλακούν πολύ περισσότερο και τα ίδια τα κράτη-μέλη. Δηλαδή, στο πλαίσιο τη αρμοδιότητα ε, που έχουν τα κράτη-μέλη να πούν ότι χρειαζόμαστε και μια ευρωπαϊκή διάσταση σε σχέση με αυτά τα ζητήματα, πέραν δηλαδή τη εθνική μα αρμοδιότητα. Και ίσω με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαμε να, πούμε, να δείξουμε στους πολίτες μας ότι σταματήστε να αμφισβητείτε το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα κοινό μέτωπο σε ορισμένα ζητήματα, ότι δηλαδή πραγματικά μιλάμε η ενιαία αναφούνη και θα πρέπει δηλαδή όταν λέμε ότι πράγματι κάτι πρέπει να γίνει στον τομέα τη απασχολήση των κοινωνικών δικαιωμάτων να προκύπτει κάτι στο τέλο μια τέτοια προσπάθεια. Να δείχνουμε ακριβώ στους ε, πολίτε μα ότι δεν του αφήνουμε μόνου μα. και μόλι τώρα συνάδελφε αναφέρθηκε στο ζήτημα τη παιδική φτώχεια. Πολλοί λένε ότι αγνοούμε αυτό το ζήτημα και όχι είναι αλήθεια και πραγματικά κάνουμε ό,τι μπορούμε και υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικά ε, ε, ε, επιχειρήματα υπέρ του ακριβώς να εμπλακούμε πιο, πιο σοβαρά και να, έχουμε ακριβώς, να δείξουμε μεγαλύτερο ενδιαφέρον για να δείξουμε ακριβώς και απέναντι στους ευρωσκεπτικιστές οι οποίοι λένε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κάνει τίποτα, ότι όχι, σταματήστε να λέτε τέτοια πράγματα. Πραγματικά έχουμε καταφέρει πολλά, έχουμε συμβάλει σε μεγάλο βαθμό και ακριβώς με αυτές τις κατευθυντήρες γραμμές της απασχόλησης. Πρόκειται δηλαδή για ε, ένα εγχείρημα το οποίο είναι τόσο ε, υπέρ τη Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και υπέρ τη Απασχόληση. Νομίζω πω με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να οδηγηθούμε σε ένα καλό αποτέλεσμα και στις επικείμενε ευρωεκλογέ. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστούμε πολύ κύριε Μαν και ευχαριστούμε και για μία ακόμα φορά τον εισηγητή τον κύριο Μητροφάνοξ. Μπορούμε να θεωρήσουμε λοιπόν ότι εγκρίνουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής χωρίς δηλαδή τροπολογίες στο πλαίσιο της απλουστευμένης διαδικασίας ε, του κανόνα 50, παράγραφος 1 του καταστατικού μας. Δεν βλέπω να υπάρχουν ε, αντιρρήσεις. Καλώς. Και βέβαια, αν υπάρχει κάποιο εκπρόσωπο από την πλευρά τη Γενική Διεύθυνση Απασχόληση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μπορεί να πάρει το λόγο. Παρακαλώ. Thank you, Chair. Το πρόεδρε. Ευχαριστώ που δίνετε το λόγο στην Επιτροπή. Θα είμαι πολύ σύντομο. Θα θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε και την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την υποστήριξή σας, για τις κατευθυντήριες αφρές. Από... Πέρσι σου λέμε το θέμα, τελικά εγκρίθηκαν και εμείς εγκρίνουμε τη διαδικασία fast track την οποία προβλέψατε για να εγκριθεί έγκαιρα η έκθεση αυτή. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Φτάσαμε στο σημείο 7 της ημερησίας διάταξης, η προσεχή συνεδριάσεις. Η επόμενη συνεδρίαση θα λάβει χώρα το πρωί της Δευτέρας Απριλίου. Έτσι. Βλέπω να, λένε, να λέει το μα. Ελπίζω όχι πριν από τι 9 το πρωί. Εν πάση περιπτώσει θα επιβεβαιωθεί. Και ελπίζω ότι θα σας ξαναδώ Όλους τις 2 Απριλίου. Δεν είναι Πρωταπριλιά, 2 Απριλίου είπα. Θα σας ξαναδώ λοιπόν. Σας ευχαριστώ που είστε παρόντες. Παρόλο που είμαστε πάρα πολύ λίγοι, ήταν σημαντική η συνεδρίαση. Και σας ευχαριστώ. Πήραμε αποφάσεις σημαντικές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για τις δυνατότητες που έχουμε να έχουμε θετικά επιχειρήματα για όλα αυτά τα θέματα όταν θα συναντήσουμε τους ψηφοφόρους μας για τις επόμενες εποχές. Ευχαριστώ. Γεια σας. Σας ξαναδώ και πάλι στις 2